και να περάσουν μετά στις ανακοινώσεις για τη θέση του Συμβουλίου πρώτη ανάγνωση για τις περιορισμούς θορύβους στους αερολιμένες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θέση του Συμβουλίου ανακοινώθηκε επίσημα στην Ολομέλεια τη Δευτέρα Απριλίου. Ο, το 63 του κανονισμού απαιτεί η θέση του Συμβουλίου να τεθεί σαν πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης υπεύθυνη καθήλυν επιτροπής την ε, πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία μετά την ανακοίνωσή της. Ο εισηγητής προτείνει την υιοθέτηση ε, της συγκεκριμένης θέσης χωρίς τροπολογίες. Τα μέλη κατέθεσαν 16 τροπολογίες, ε, θα ακολουθήσει η ψηφοφορία. Έπρεπε όμως να κάνω την τυπική ανακοίνωση διότι θα γίνει ανακοίνωση και στην Ολομέλεια. Έχουμε και την έγκριση των πρακτικών της 17ης και 18ης, 21ης ε, Μαρτίου και 1ης Απριλίου. Δεκτά. Περνάω λοιπόν στη μείωση του θορύβου, δεύτερη ανάγνωση. Η συγητής είναι ο κύριος Λάιχτφεϊντ. Θα περάσουμε στην ψηφοφορία, δοκιμάζομαι το μηχανισμό ψήφου, άρχεται η ψηφοφορία. Has everybody voted? No. Ψηφίσατε όλοι. Ποιο ψηφίζει με την πιστοτική του εδώ. Πέρα της ψηφοφορία. Εντάξει. Και ο κύριος Γκρός δεν έχει την κάρτα του. Περνάμε τώρα στις 15 τροπολογίες τις οποίες θα ψηφίσουμε ομαδών. Τι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Είναι ασυνήθιστο, Μάικλ, που το λέω στη μέση της ψηφοφορίας, αλλά στην ουσία τελειώνουμε όπως ξεκινήσαμε. Τελική ψήφος. Α, για μια στιγμή. 14, απολογία 14, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίφθη. Ηλεκτρονικός έλεγχος ζητά ένας βουλευτής. Λοιπόν το 15 διαγράφει Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 16 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 5 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Περνάμε τώρα στην τελική ψήφο, άρχεται η ψηφοφορία. As everybody voted, the vote is... Ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. 19 υπέρ, 4 κατά. Καμία αποχή. Δεκτή. <clears throat> Συγχαρητήρια στον κύριο Λάιφεντ. Επόμενο θέμα. καταληκτικές παρατηρήσεις από τον Πρόεδρο στο τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου. Οι συνάδελφοι θα έχουν ίσως διαβάσει ήδη. Το βιβλιαράκι το οποίο βάλαμε στα καζιέ σας. Βλέπω εδώ ότι έχει και εκπληκτικές φωτογραφίες, ιδιαίτερα ευηδών μελών της Επιτροπής μας. Μπορείτε αντίγραφα περισσότερα να πάρετε από τη γραμματεία εφόσον τα έχετε ανάγκη. Αυτή τη φορά είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έχουμε βάλει φωτογραφίες μαζί με τις εκθέσεις του κάθε εισηγητή και αυτό ήταν μια καλή ιδέα, όπως είχε άλλωστε ζητηθεί. Και είναι και καλά σχεδιασμένο. Λοιπόν θα ήθελα να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις για να κλείσουμε αν μου επιτρέπετε ως πρόεδρο. Τερματίζονται οι δραστηριότητες μας σαν Κοινοβουλευτική Επιτροπή εκτός από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα. Ήταν μια ιδιαίτερα βεβαρημένη πλούσια όμως ε, κοινοβουλευτική περίοδος, ιδιαίτερα το δεύτερο ήμιση της κοινοβουλευτικής περίοδου. Το έχουμε ξαναπεί αυτή, ιδιαίτερα σε σχέση με την νομοθετική δραστηριότητα η οποία καθυστέρησε. Ήμασταν πολύ δραστήριοι λοιπόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη σκληρή σας δουλειά κατά τη διάρκεια της προηγούμενης πενταετίας και δεν συμπεριλαμβάνω μόνο τα πλήρη μέλη αλλά και τους αναπληρωτές. Είχαμε πάρα πολλούς αναπληρωτές ιδιαίτερων δραστήριους. Όταν βλέπει κανείς το τι έχουμε κάνει τα τελευταία πέντε χρόνια διαπιστώνει ότι έχουμε κάνει αρκετά τα οποία ωφελούν τις μεταφορές στο εσωτερικό της Ένωσης. Υπάρχουν πολλά που μένει να γίνουν βέβαια έτσι ώστε τα συστήματα να γίνουν πιο ολοκληρωμένα από ό,τι σήμερα. Αλλά θέλει χρόνο αυτό, πρέπει να πείσουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν τις απαιτούμενες αλλαγές. Θα ήθελα να εκφράσω τα ευχαριστήριά μου επίσης στο προσωπικό της Επιτροπής, στην Επιτροπή Τουρισμού και Μεταφορών και αυτούς που ήταν συνεχώς μαζί μας και αυτούς οι οποίοι ήρθαν και μετά πήγαν σε άλλα τμήματα. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τους υπαλλήλους των βουλευτών οι οποίοι πράγματι ε, διασφάλισαν τους κλητήρες φυσικά που μας έδωσαν χιλιάδες έγγραφα έτσι ώστε τα έγγραφα να είναι έτοιμα, αλλά κυρίως το μαγικό έγγραφο να είναι έτοιμο για να υπογράψουμε όταν μπαίνουμε στην αίθουσα. Και θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τη Διεμηνία. Εγώ είμαι κλασικό παράδειγμα α, βουλευτή χωρίς τους οποίους δεν θα μπορούσαν να κάνω τίποτα. Πολλές φορές Λέμε ότι ο πρόεδρος δεν μιλάει καλά αγγλικά, αλλά δεν μιλάει και καμιά άλλη γλώσσα καλά. Πρέπει να το υπογραμμίσω αυτό. Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά την οποία κάνουν. Κάθονται πολλές φορές τρει ώρες, τρεις ώρες, τρεις ή μισή ώρες μέσα στον θαλαμίσκο τους, διευρυνεύοντας αυτά τα οποία λέμε. Σε τομείς οι οποίοι είναι αρκετά τεχνικοί θα έλεγα. Το κάνουν αυτό με επαγγελματισμό και μεγάλη αποτελεσματικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους διευμηνείς σε όλες τις καμπίνες για τη σκληρή τους δουλειά τα προηγούμενα πέντε χρόνια και εμείς θα τα αποδίδουμε. So now we, we move on. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ο Μάθιου και εγώ κάποια στιγμή θα κληθούμε να δώσουμε τη μαρτυρία μας από τη νέα Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Όσοι ζητάτε να επανεκλεγείτε, σκοπεύετε να επανεκλεγείτε, καλή τύχη. Όσοι αποσύρεστε, σας εύχομαι μια μακρά και ευτυχή περίοδο συνταξιοδότησης. Ελπίζω να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε. Προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί σε καθημερινή βάση Thank you as well. θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο ο οποίος ήταν κολλητός μας όλα αυτά τα χρόνια. Τον ευχαριστώ για την βοήθειά του και επίσης και τους υπαλλήλους των πολιτικών ομάδων που συνεχώς μας τροφοδοτούν σε έγγραφα και μας οδηγούν πάντα στον σωστό δρόμο. Θέλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους των γραφείων μας που μας στήριξαν σε μόνιμη βάση έτσι ώστε να μην χάσουμε το δρόμο μας και να κάνουμε καλή δουλειά. Συνεχίζουμε όμως τώρα. Εύχομαι σε όλους και στην Επιτροπή λοιπόν ό,τι καλύτερο και σε εσά προσωπικά και στο προσωπικό σας. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα είναι η επόμενη κοινοβουλευτική επίτροπος τόσο καλή όσο η παρούσα. Και αυτό γιατί αυτή η επιτροπή είναι απολύτως η καλύτερη επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο λόγος για τον οποίο είναι είναι λόγω του Προέδρου λέει ο Μάικλ είναι λόγω της δικής σας παρουσίας. Εσείς τα μέλη καταστήσατε την Επιτροπή αυτή την καλύτερη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας και εύχομαι καλή τύχη σε ό,τι κάνετε από εδώ και πέρα. Και καλά ταξίδια στο μέλλον. Ευχαριστώ. I have to announce the date and time of the next meeting. Πρέπει να ανακοινώσω τι 7 Ιουλίου στι 3 ε, θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση. Μάτιο Γκρός. Ναι. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και εγώ, αλλά να ευχαριστήσω και όλους και σένα συγκεκριμένα διότι ε, το γεγονός ότι εξελίχθηκαν οι εργασίες της Επιτροπής ε, με τον τρόπο που εξελίχθηκαν ε, οφείλεται και στην, στη μορφή της συνεργασίας μας. Χθες και νομίζω ότι ήταν μια πολύ ευχάριστη ευκαιρία είχα την ευκαιρία να πω ότι στην Επιτροπή μας είναι, γνωρίζουμε ότι η οικοδόμηση γεφυρών είναι κάτι πολύ σημαντικό και δεν προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό μόνο στην Ευρώπη. Νομίζω το καταφέραμε και εδώ εντός της Επιτροπής. Χτίσαμε δηλαδή σε πολλά σημεία γέφυρες μεταξύ διαφορετικών γνωμών και παρότι δεν καταφέραμε να, κάνουμε όλα όσα θέλαμε μεταξύ των ομάδων, νομίζω όμως ότι σε ουσιώδη σημεία και σε ουσιώδη θέματα καταφέραμε να επιτύχουμε ουσιώδης στόχους. Να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μου, τον Βάλτα Γκέρτς. Πρόκειται, το έγγραφο αυτό είναι μια, η, η ολοκλήρωση ενός πολύ σημαντικού έργου και χθες μίλησα με την ε, προκάτοχό σου που μου είπε ότι είναι ευτυχία, είναι ευτυχία στο γεγονός ότι η γραμματεία ε, διαθέτει τόσους ικανούς ανθρώπους, ίσως δεν διαθέτει τον απαραίτητο χρόνο, αλλά διαθέτει ανθρώπους που γνωρίζουν την ε, υπόθεση. Και το ίδιο ισχύει και για, τους, ε, για τις ομάδες και όποιος έχει υποβάλει εκθέσεις ξέρει ότι η συνεργασία είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Για τους ε, μεταφραστές και το προσωπικό θα ήθελα και εγώ να πω ε, ιδιαίτερα ως Γερμανός ε, ξέρω ότι είναι ένα πολύ δύσκολο έργο διότι υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές της γερμανικής γλώσσας, βελγικά, λουξουμβουριανά Στην, στην αγγλική γλώσσα υπάρχει μόνο μία εκδοχή αυτής της γλώσσας αλλά στην ε, καμπίνα οι διερμηνείς έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορα είδη γερμανικών αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, η επιτυχία των εργασιών μας ε, ε, οφείλεται και σε εκείνους. Και τέλος, ασχοληθήκαμε με 180 προτάσεις εδώ στην Επιτροπή και νομίζω ότι τις υπερψηφίζαμε με μεγάλη πλειοψηφία τις περισσότερες φορές. Όχι γιατί το τέλος ήταν τόσο κακό, αλλά το αντίθετο, επειδή το τέλος ήταν καλό. Και με 50 νομοθετικές προτάσεις θα ήθελα να ε, εκφράσω τις ευχαριστίες μου μεν και στην Επιτροπή αλλά θα ήθελα επίσης να πω ε, ότι πρέπει να παραμείνει στις επάλξεις για τις ε, μεταφορές διότι ε, γνωρίζουμε ότι πάρα πολλοί άλλοι το, τομείς θέλουν να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα που ασχολούμαστε εδώ αλλά εμείς είμαστε οι αρμόδιοι και γι' αυτό θα ήθελα να ευχηθώ ε, και στο μέλλον οι μεταφορές και η κινητικότητα να παραμείνει αυτόνομος τομέας και όχι υποτομέας άλλων τομέων. Και τέλος να πω κάτι που έμαθα από σένα. Ε, θα ήθελα να πω αυτό που έλεγες και εσύ πολλές φορές στο τέλος. Ελπίζω όλοι να είστε ευτυχισμένοι και εγώ μπορώ σε κάθε περίπτωση να σας πω ότι ήμουν ευτυχισμένος εδώ σε αυτή την Επιτροπή ως Γερμανός. Ευχαριστώ. Thank you Matthew. Said. I've got Said and <clears throat> Michael. Yeah, Michael. Ευχαριστώ. Θα ήθελα με τη σειρά μου και εγώ να απευθύνω τις ευχαριστίες μου προς όλους όσους συνέβαλαν στα παρασκήνια στην ε, επιτυχή απόλυξη των κοινοβουλευτικών μας εργασιών. Ευχαριστώ όλες τις κατηγορίες του προσωπικού, ευχαριστώ τους διερμηνείς, ευχαριστώ το προσωπικό νομίζω ότι είναι μεγάλη συμβολή τους ως προς τα τελικά αποτελέσματα των εργασιών μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς, Πρόεδρε. Ε, το βράδυ ήδη όταν συναντηθήκαμε είπα αρκετά πράγματα. Νομίζω και το επαναλαμβάνω ότι είστε από τους πιο πεπειραμένους ε, προέδρους ε, και όταν λέω πεπειραμένος το εννοώ ε, από πολλές πλευρές διότι κατέχετε πλήρως τον κλάδο για τον οποίο είστε αρμόδιος τα 20-30 τελευταία χρόνια ουσιαστικά συμμετείχατε σχεδόν σε όλους τους φακέλους ε, που πραγματεύτηκε η Επιτροπή Μεταφορών. Έχουμε όλοι έντονα την εντύπωση ότι ήσασταν ιδιαίτερα προσιλωμένος, ε, ήταν ισχυρότατη η δέσμευση που επιδείξατε για να έχουμε μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία χάρη στις εργασίες μας. Όπως είπατε θα συναντηθούμε ενδεχομένως ε, σε κάποιο άλλο πλαίσιο. Και ίσως ε, βρεθείτε εσείς στη θέση στην οποία βάζατε ε, τους ε, προσκεκλημένους μας, δηλαδή ενώπιον ενός αυστηρού αλλά και ακριβοδίκαιου Προέδρου κατά τη διάρκεια των της εξέτασης των διαφορών ζητημάτων. Ε, υπάρχουν πολλοί βουλευτές που δεν θα επιστρέψουν, όπως εσείς, η ε, Ματιέ. Ε, ένα δε χαρακτηριστικό της Επιτροπής μας είναι ότι επικρατούσε ένα επικοδομητικό πνεύμα που παρά τις διαστάσεις απόψεων μας επέτρεπε να καταλήγουμε κάθε φορά σε συνενετικές θέσεις και σε ένα αποτέλεσμα που οδηγούσε σε βήματα πρόοδου κάθε φορά. Έχουμε ε, συγκεκριμένα αποτελέσματα, απτά αποτελέσματα στο ενεργητικό μας και αυτό θα έχει ιδιαίτερη σημασία στην προεκλογική εκστρατεία. Ευελπιστώ ότι θα επανεκλεγούν όλοι όσοι το επιθυμούν και για τους υπολείπους ε, καλή τύχη στο νέο κεφάλαιο της ζωής σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συναδέλφους. Πραγματικά ήταν πολύ ευχάριστη η δουλειά εδώ ε, στο, στην Επιτροπή με τους ε, συνεργάτες, με τη Γραμματεία, ακόμα και με τους εκπροσώπους της Κομισιόν. Έχουμε σήμερα εδώ. Ναι, και φυσικά θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς και να ευχαριστήσω και σένα προσωπικά, Μπράιαν. Πραγματικά ήταν πολύ κρίμα που χθες δεν μπόρεσα να έρθω, θα ξανά, έχω το σκοπό όμως να ξανάρθω. Ε, ε, είμαι, στην, στην, είμαι υποψήφια στη Γερμανία, ε, γι' αυτό και έλειπα χθες και θα είμαι και στην επόμενη ψηφοφορία. Γι' αυτό δεν θα μιλήσω πολύ σήμερα. Πραγματικά ήταν πολύ ευχάριστη η δουλειά εδώ και το έγραψα και στο βιβλίο ότι Μπράιαν ε, δεν ξέρω βεβαίω όλου του πρόεδρου τη επιτροπή, αλλά ήμουν και σε, έχω υπάρξει μέλο και σε επιτροπή άλλων κοινοβουλίων. Εσένα θα έδινα το, το Όσκαρ, όχι γιατί είσαι απλά ε, καλός άνθρωπος, αλλά γιατί είσαι και πολύ δίκαιος πρόεδρος. Κάποιες φορές είχαμε την αίσθηση ε, ότι ενδεχομένως να μεροληπτείς, αλλά εγώ τις περισσότερες φορές στην αρχή δεν ήξερα καν σε ποια πολιτική ομάδα ανήκεις, γιατί, δεν, γιατί ακριβώς ήσουν τόσο δίκαιος. Βεβαίω, όλοι έχουμε τι πολιτικέ μα απόψει, αλλά όταν κάθεται κανεί εκεί μπροστά, ε, έχει πάλι, εξακολουθεί να έχει μια άποψη, αλλά ε, πρέπει να διασφαλίζει ότι όλοι ε, έχουν ε, το δικαίωμα να τοποθετούν. Και νομίζω ότι εσύ το έκανε πολύ καλά, διότι αυτό είναι και η ουσία τη δημοκρασία, να καταμερίζει κανεί δηλαδή από τη δική σου θέση και τον χρόνο δίκαια. Και δυστυχώ πρέπει να φύγω αλλά νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε και στην ε, Ολομέλεια και ελπίζω να δω και στην επόμενη θητεία πάρα πολλούς από τα παλιά μέλη. Και χαίρομαι πάρα πολύ με αυτή την προοπτική. Well, Σε ευχαριστώ. Αν δεν ξέρουν οι επισκέπτες τους μετά από όλα αυτά που ακούσανε, σοσιαλδημοκράτης είμαι. <laughs> Αλλά και εκεί πέρα λίγο, πώ να πω, περιθωριακό είμαι, μπορεί κάποιο να το αμφισβητήσει ότι ανήκω στου Ελληνικοκράτε Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω, Μπάιαν, εσένα προσωπικά και για το εξαιρετικό βρετανικό σου χιούμορ Ευχαριστώ και τους ε, συναδέλφους για τις συνεισφορές τους. Ακόμη και αν δεν είχαμε πάντοτε την ίδια άποψη, αυτό είναι σαφές. Διότι η δική μου ομάδα πολλές φορές ιτάται στις ψηφοφορίες, αλλά σε σύγκριση με άλλα κοινοβούλια νομίζω ότι είχαμε πολύ ουσιώδεις αντιπαραθέσεις και αυτό είναι σημαντικό. Να μπορεί δηλαδή κανείς και επιστημονικά, τεχνικά να αντιπαρατίθεται και παρόλα αυτά να θεσπίζει μια καλή στρατηγική. Επίσης εκτίμησα ιδιαίτερα το γεγονός, ήμουνα και σε άλλες επιτροπές κατά καιρούς, ότι οι ψηφοφορίες, οι διαδικασίες εδώ σε αυτή την επιτροπή εξελίσσονταν πάντοτε ομαλά, δεν υπήρχε κανένα σημείο κριτικής δεν είναι αυτονόητο αυτό για άλλες επιτροπές. Και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους ε, μεταφραστές διότι ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών ε, τα... οι δυσκολίες είναι μεγάλες. Υπάρχει ειδικό λεξιλόγιο και μάλιστα πάρα πολλές γλώσσες που είναι πολύ δύσκολο να αποδίδονται όλες αυτές οι μικροδιαφορές. Να ευχαριστήσω λοιπόν σίγουρα τους ε, μεταφραστές και βεβαίως και τη γραμματεία που επιτέλεσε πολύ σημαντικό έργο. Εγώ δεν θα επανέλθω στο κοινοβούλιο, αλλά ενδεχομένως ε, θα με ξαναδείτε σε ακτιβίστρια, σε πρωτοβουλίες, κάποια από εσάς, διότι τα, τις τελευταίες φορές υπήρχαν δύο αλπίνο, σήμερα είναι μόνο μία αλπίνο, την, την επόμενη φορά μάλλον δεν θα υπάρχει κανείς, ε, οπότε θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην ξεχάσετε τις Άλπεις. Είναι ένα σημαντικός τομέας για τις ε, μεταφορές. Γι' αυτό κατά καιρού θα σας στέλνω κάποιο γράμμα για να σας επιθυμίζω αυτήν την επιθυμία μου και μπορεί και να έρχομαι από καιρούς καιρών ακριβώς για να τονίζω αυτήν την επιθυμία μου διότι η ε, Άλπης είναι και ένα μέτρο ελέγχου για την ε, πολιτική μεταφορών ότι δεν λειτουργεί εκεί, δεν θα λειτουργήσει μακροπρόθεσμα ούτε σε άλλα εδάφη οπότε σας ε, προειδοποιώ ότι θα επανέρχομαι συχνά για να σας υπενθυμίζω τις Άλπης ακριβώς γιατί δεν θα έχουμε μάλλον στην επόμενη θητεία κανέναν που να υπερασπίζεται το συγκεκριμένο θέμα αλλά Ενδεχομένως επίσης να σας ε, ε, συναντήσω στο Τυρόλο σε, σε σκι, σε διακοπές σκι. Εγώ θα σας κάνω ε, με πολύ μεγάλη μου χαρά ένα μάθημα σκι, αν θέλετε, όποιος θέλει. Σε κάθε περίπτωση καλή τύχη σε όλους όσους συνεργάστηκαν εδώ μαζί μας. Και Brian, καλή τύχη σε σένα προσωπικά. τώρα που μεταβαίνεις από, τον, ε, από τους ιδεοδρόμους στη θάλασσα. Είναι δύσκολος ο τομέας αυτός, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρεις. Well, thank you all and... Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Καλή επιτυχία σε όλους και εγώ εύχομαι. Ε, Βεβαίω ε, δεν θα ήταν σωστό ο αποχαιρετισμό από πλευρά ενό Μπράιαν Σίμψον αν δεν μιλούσα και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα προειδοποιώ λοιπόν, όπω σα έλεγα και νωρίτερα, δεν μιλώ μόνο για τη γαμαδέλτα Move του Φιλ. Γενικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πραγματικά, εν πάση περιπτώσει, ε, να παρακολουθείτε στενά την DigiCom <laughs> γιατί θα ε, θα γίνει χαμός ε, αν δεν τους ελέγχετε στενά. Ε, εγώ φεύγω πάντως πατώντας την, τον παλιό μου εχθρό, την DigiComp. Ο Μπλερ στην τελευταία ώρα ερωτήσεων στη Βουλή είπε το εξή διάσημο τέρμα. Τελείωσαν όλα. It's all finished. Έτσι κλείνω και εγώ. Γεια σας.